όποια Επεξηγήσεις ε, ε, ψήφου. Πρώτα απ' όλα για την έκθεση Ριέρα Μαντουρέλ, συνάδελφος Χένεν. Εδώ παρόν. Yes, please, you have the floor. Έχετε τον λόγο. The field of το θέμα της ίσης αμοιβή και της ισότητας των φύλων είναι το υπέρτατο παράδειγμα εντός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικής δραστηριοποίησης. Ένα λέει συνθήκη ακτιβισμό, ένα λέει συνθήκη και κάτι άλλο γίνεται. Μία πρόταση του θέματος είναι, θα έλεγε κανείς, ότι είναι πολύ εύληπτη οι άνδρες και οι γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο για ίση εργαστήρια. Όμως έχουν υπάρξει ε, πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις, ας πούμε η, τη Σαμπένα, του Guardian κλπ, που έχουν οδηγήσει σε διαφορές και στις συντάξεις κλπ. Και το εργασία ίσης αξίας πώς θα αξιολογηθεί δεν είναι βέβαιο. Τι τι σημαίνει για ένα εργοστάσιο η, διαθεση, η ύπαρξη ε, κατάλληλων υποψηφίων. Το θέμα είναι ότι τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι έχουν υπογράψει μία συνθήκη την οποία διαπιστώνουν ότι τα δικαστήρια ερμηνεύουν διαφορετικά χωρίς να ερωτηθούν αν αυτό επρόκειτο να, αυτό είχαν σκοπό να ε, ψηφίσουν οι νομοθέτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλέ επί του ιδίου θέματος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν συμφωνώ με την έκθεση αυτή. Όχι διότι είμαι κατά της ίσης μεταχείρισης ε, ανδρών και γυναικών στο χώρο της δουλειάς, αλλά επειδή έχει, μιλάμε για τρέλα της πολιτικής ορθότητας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς μπορεί κανείς να αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης. Ζούμε σε χώρες που στηρίζονται στο κράτος δικαίου και δεν πιστεύω ότι πρέπει να αντιστραφεί το βάρος της αποδείξεως υπάρχει υποχρέωση κάθε χρόνο να υπάρχει ε, επιχειρηματικό σχέδιο για την ε, ισότητα των φύλων. Και αυτό είναι φοβερό. Αναγκάζουμε τις ε, επιχειρήσεις να κάνουν περιττές διαδικασίες επί τη βάση αρχών που είναι αποδεκτές σε όλους και οι οποίε όμως δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν στην πράξη. Πώς είναι δυνατόν να επιβάλλουμε σε μια εταιρεία να προσλαμβάνει ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών κάθε χρόνο. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Μέση Ανατολής και τη Λόριδα της Γάζας, έχουν δηλώσει πολλοί ομιλητές. Κύριος Γκρέγκερ. Δεν τον βλέπω να... στην αίθουσα. Κυρία Μπικίνη. Πρόεδρε, υπερψήφισα το ψήφισμα για την κατάσταση στη Γάζα, διότι πολλά πράγματα που είναι σημαντικά για τους Λιθουανούς περιλαμβάνονται στο κείμενο του ψηφίσματος. Το πιο σημαντικό είναι η συμφωνία για την εκεχηρία. Τα στατιστικά στοιχεία που έδωσαν χτες τα μέσα ενημέρωσης είναι εντυπωσιακά. Ε, πάνω από χίλιοι νεκροί πλέον, ε, χιλιάδες τραυματίες μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά. Ω μέλο τη της Υποεπιτροπή Δικαιωμάτων των Ανθρώπων, ενδιαφέρουμε ιδιαίτερα για την ανθρωπιστική κατάσταση και την παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο στην ανθρωπιστική βοήθεια που θα πρέπει να φτάνει αυτού που την χρειάζονται, κατά βάση τον άμαχο πληθυσμό. Καλωσορίζω το ψήφισμα από πλευρά Κοινοβουλίου. Πραγματικά ε, είναι αναγκαίο και δεν έπρεπε το Κοινοβούλιο να σιωπά όταν ο κόσμο σκοτώνεται. Ευχαριστώ κύριε Μακίνε. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να χαιρετίζουμε το ψήφισμα για τη Γάζα το οποίο φυσικά το χαιρετίζω γιατί τέτοιου είδους ε, λόγια δεν ακούστηκαν παρά τις φωνές ε, των πληγωμένων και αυτών που δολοφονούνται στην περιοχή. Σήμερα όμως θα πρέπει να γίνουν περισσότερες κινήσεις προς κατάπαυση του πυρός. Αυτό θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτο. Υπό την έννοια αυτή υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Αιγύπτου να επιτύχει κατάπαυση του πυρός και παρότι η Αίγυπτος μπορεί να επηρεάσει τη Χαμάς όσον αφορά το Ισραήλ την επιρροή την έχει οι Ηνωμένε Πολιτείε Ελπίζω ότι το ψήφισμα το οποίο ε, υποστηρίχθηκε ε, από το σώμα σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία ε, χωρίς να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια και χωρίς κατάπαυση του πυρός δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ κύριο Χάναν. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα χάρηκα που είδα για το ότι δεν τιμωρήθηκαν οι συνάδελφοι που σήκωσαν τα πλακάτ ε, εδώ πέρα. Ελπίζω λοιπόν να δημιουργήθηκε ένα προηγούμενο, δηλαδή μπορεί κάποιο ειρηνικά να εκφράσει απόψη εκτό βεβαίω όταν μιλάμε για το δημοψήφισμα. Όπω και όλοι οι υπόλοιποι βεβαίω, έτσι και εγώ νιώθω φρίκι για αυτά τα οποία συνέβαιναν και αυτοί οι οποίοι θα χάσουν δεν είναι η μία ή η άλλη πλευρά, αλλά οι άνθρωποι σε ολόκληρη την περιοχή. Οι οικογένειε στην Γάζα προσπαθούν να αναθρέψουν τα παιδιά τους και βεβαίω ε, με φρίκι βλέπουν το τι συμβαίνει. Είναι οι Ισραηλινοί που αντιλαμβάνονται ότι μία μέρα θα έχουν μια ανεξάρτητη Παλαιστίνη γείτονα και με τέτοιες δράσεις βεβαίως δεν θα είναι καθόλου φιλικός γείτονας. Αλλά αυτές οι φωνές δεν ακούγονται. Επίσης δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοεί με την αναλογικότητα το ψήφισμα. Θα ήταν ε, ικανοποιημένοι, δηλαδή όσοι ασκούν κριτική στο Ισραήλ, εάν είχε πέσει ένας εξίσου μεγάλος αριθμός ε, βλημάτων ε, στα Ισραηλινά χωριά όπως αυτά τα οποία έπεσαν στην Γάζα. Σας ευχαριστώ κύριος Πόσελτ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Τσεχίας και Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Σφάρτσεμπερ και την κυρία Φερέρο Βάλτνερ για αυτά τα οποία μας είπαν ε, χτες και για την σημερινή σχεδόν ομόφωνη πλειοψηφία. Θεωρώ πως επιδεικνύουμε μία αποφασιστικότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μπορούμε να επιτύχουμε και κάτι και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την γραμμή. Τα στοιχεία είναι σαφή τα βασικά. Ναι, υποστηρίζουμε το δικαίωμα ύπαρξη Ισραήλ, όχι στον πόλεμο και στην αιματοχυσία, όχι στις ρακέτες της Χαμάς, όχι στο τρομοκρατικό σύστημα της Χαμάς και κάτι το οποίο είναι εξίσου ουσιαστικό, χρειαζόμαστε διαπραγματεύσει για τα επίμαχα σημεία και του ζητήματος των επίκων που είναι το ζήτημα που είναι πυρήνα εδώ πέρα δίπλα με τον απαράδεκτη τρομοκρατία της ε, Χαμάς. Οπότε θεωρώ πως αποστολή μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να κινήσουμε αυτή την υπόθεση με ενεργεία και αφασιστικότητα και να μην γινόμαστε πάλι μια διχασμένη λέσχη συζητήσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάκουλα για την έκθεση αυτή τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή αυτή και άμεση εκεχηρία. Για να πετύχουμε εκεχηρία ωστόσο πρέπει να αγωνιστούμε ούτως ώστε να αφαιρεθούν τα όπλα από την Χαμάς και πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε με πιο εμφαντικό τρόπο στο ψήφισμα. Καταλαβαίνω ωστόσο ότι όταν ετοιμάζουμε συμβιβαστικά κείμενα μεταξύ διαφόρων πολιτικών ομάδων, δύσκολο μπορεί να πετύχει κανεί όλα όσα θέλει. Πρέπει ω Ευρωπαίοι να λειτουργούμε αντικειμενικά. Σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία και πρέπει να, αντιτιθέμεθα στην τρομοκρατία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Επίση, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό το, όλο αυτό το πρόβλημα ξεκίνησε λόγω των δημοκρατικών επιθέσεων. Και του δημοκράτε αυτού πρέπει να του ξεφορτωθούμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που το Κοινοβούλιο μπόρεσε να εγκρίνει το ψήφισμα με τόσο εντυπωσιακή πλειοψηφία εμείς και εγώ προσωπικά το υποστηρίξαμε γιατί θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη θέση και να ε, στηρίζεται σε κοινέ απόψεις παρότι η θέση δεν αντιπροσωπεύει 100% την ε, άποψη της σοσιαλιστικής ομάδας. Επαναλαμβάνω ότι η σοσιαλιστική ομάδα εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας γιατί η στρατιωτική κλιμάκωση έχει διοδηγήσει σε σε πολλούς θανάτους μεταξύ των οποίων αμάχουν και παιδιά. Έχουν πληγεί επανειλημμένως ε, άμαχοι. Επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχει ε, είναι απαραίτητο οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ θα πρέπει να στηρίζονται στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε θέματα ανθρωπιστικού δικαίου, την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και να γίνει πλήρης εφαρμογή της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης πιελό. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούλινγκ θα έχει δει στο λόγο. Μισό λεπτό κύριε Λούλινγκ. Διαδικαστικό για την έκθεση Μαντουρέλ ζητήσατε. Ωστόσο, τα διαδικαστικά αφορούν μόνο επί του προσωπικού. Προτείνω να, κάνει, να πείτε αυτό που θέλετε μέσω τη επεξήγηση ψήφου. Ακριβώ, σωστά. Και γι' αυτό το λόγο έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί σε κάποια προφορική ε, επεξήγηση ψήφου ενό συναδέλφου αναφέρθηκαν απίθανα πράγματα. Είπε δηλαδή ότι το ψήφισμα περιλαμβάνει πράγματα που είναι ανακριβή δεν υπάρχει υποχρέωση των εργοδοτών να παίρνουν έναν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών. Αποσύραμε τις υποχρεώσεις, όλες τις υποχρεώσεις από την έκθεση έτσι όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Υποβάλαμε ένα κοινό ψήφισμα και ελπίζω ο συνάδελφος αυτός να μην είναι αντίθετος με το γεγονός ότι ζητάμε υπογραμμίζουμε την ανάγκη να ενθαρρυνθεί ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ούτως ώστε να εφαρμόζεται η αρχή και αυτή και ότι δεν είναι κόντρα στο ότι ζητούμε από τα κρατημέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να προσφέρουν τακτικά στους εργοδότες και σε τους εκπροσώπους τους πληροφορίες ε, για τον σεβασμό της αρχής της ισότητας και ελπίζουμε να μην είναι κόντρα στο ότι ζητούμε τα κρατημέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να παρέχουν τακτικά πληροφορίες. Ό,τι κατέκρινε λοιπόν δεν περιλαμβάνονται πλέον στο ψήφισμα που εγκρίναμε. Ήθελα να το πω αυτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ για την επεξήγηση ψήφου που ήταν σαφέστατη. Φτάσαμε τώρα στη δήλωση Συμβουλίου και Κομισιόν ε, για τη στρατηγική της, του Συμβουλίου απέναντι στην ε, Λευκορωσία, κυρία Αντρίκη. Υπερψήφισα το ψήφισμα κύριε Πρόεδρε για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρευκορωσία, δεδομένου ότι θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει πολύ σωστά τις αλλαγές που επήλθαν το τελευταίο εξάμεινο στη χώρα. Το ότι έχουν υπάρξει πρώτες ενδείξεις φυσικά δεν συνεπάγεται ότι έχει γίνει σοβαρή πρόοδος Χαιρόμαστε όμως ιδιαίτερα για οποιαδήποτε αλλαγή όπως ε, απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, περιορισμό των ε, απαγορεύσεων στη ελευθερία του τύπου κλπ. Αυτά είναι πολύ θετικές ενδείξεις και σήμερα θέλω να διαβεβαιώσω ότι πλέον πιστεύουμε ότι έφτασε η στιγμή να πάει μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκορωσία όπως λέει και το ε, ψήφισμά μας. Όταν η Λευκορωσία θα μπορέσει να εποφεληθεί από την ε, πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απέχει πολύ. Πρέπει να μην σταματήσουμε όμως ενδιάμεσα. Πρόεδρε, καταψήφισα το ψήφισμα παρά το ότι περιλαμβάνονται οι αξιόπιστα και ενδιαφέροντα στοιχεία ισορροπημένα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι για να διατηρήσουμε ένα καθεστώς κυρώσεων έναντι της ε, Λευκορωσίας. Από την άποψη των οικονομικών, πολιτικών και θρησκευτικών ελευθεριών η χώρα αυτή είναι μια χώρα που τήρησε σχεδόν πλήρως τα κριτήρια ελευθερίας που πιστεύουμε ότι, στα οποία πιστεύουμε και εμείς. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε πραγματικές σχέσεις με την Λευκορωσία ούτως ώστε να ενταχθεί η χώρα αυτή στην Ευρώπη πλήρως. Ιδιαίτερα στην φάση αυτή όπου χρειάζεται να ξεκινήσουμε επαφές και με τη Ρωσία. Η Λευκορωσία μπορεί να αποτελέσει καλή γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Θεωρώ δε ότι αντί να απειλούμε τη χώρα με κυρώσεις πρέπει να ξεκινήσουμε έναν καρποφόρο διάλογο και μια καρποφόρα σχέση με τη χώρα αυτή. Δεν υπάρχουν άλλοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Διακόπτουμε λοιπόν την συνεδρίαση. Θα ξεκινήσουμε εκ νέου στι 3 για τις συζητήσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, ε, κράτους δικαίου κλπ. Καλή σα όρεξη.